Ε, καθίστε παρακαλώ, αρχίζουμε. Είμαστε στο σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο για την απογευματινή συνεδρίαση, παρουσίαση ε, της ε, κοινή ανακοίνωσης ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Λατινική Αμερική και Καραϊβική ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα κοινό μέλλον. Βεβαίως, όχι όλο μας το μέλλον, τα εμπορικά θέματα. σε σχέση με τις ε, εμπορικές συμφωνίες που συζητούμε με τη Λατινική Αμερική, Έχουμε μερικές ενισχύει ήδη με τις χώρες, κάποιες χώρες της Καραϊβικής και χρειάζεται να προβληματιστούμε πιο στρατηγικά για το πώς έχει το κοινό μας μέλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το εμπόριο πάντα. Έχω εδώ δύο εμπειρογνώμονες να καλωσορίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή, ε, μάλλον την Περιπηρεσία Εξωτερική ε, δράση ο Ματία Χιόγκερσον, γνωστό και μη εξαιρετέω και η Κλάουντια Χίντερστορφερ, που θα μας κάνουν την παρουσίαση και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προοπτικές. Ματίας, 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Επιτροπή σας ε, στην πρώτη μου εμφάνιση εδώ στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς από πλευράς μας θέλουμε να συνεχίσουμε τη γόνιμη και πολύ στενή συνεργασία που είχαμε με το Κοινοβούλιο. στο θέμα μας. Είδατε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση για τη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν καλύπτει αμυγός θέματα εμπορίου. Είναι βεβαίως πολύ ευρύτερη. Αλλά σήμερα είναι γεγονός ότι το εμπόριο και οι επενδύσει αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Όταν λοιπόν ελήφθη η απόφαση αυτή να εκδοθεί η συγκεκριμένη ανακοίνωση, ήταν φυσικό και επόμενο να ε, εξεταστούν και θέματα εμπορίου. Και μάλιστα είναι σημαντικό κεφάλαιο το εμπόριο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες στην ανακοίνωση αυτή. Δεν είναι κάτι το καινούριο για σας. Βασίζονται σε ε, προτεραιότητες που είχαμε. Ευημερία, δημοκρατία, ανθεκτικότητα και ε, παγκόσμια δημοκρατική διακυβέρνηση και αποτελεσματική. και το εμπόριο είναι παντού. Παράδειγμα, ε, ε, παγκόσμια διακυβέρνηση, αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση, υπογραμμίζουμε ότι θα εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στα πολυμερή φόρα και ιδιαίτερα στον ΠΟΕ που είμαστε εταίροι και συνεργαζόμαστε και τα επόμενα χρόνια έτσι αναμένεται να γίνει. Ε, το εμπόριο λοιπόν ε, συνεισφέρει σημαντικά. Και το επόμενο θέμα της ανθεκτικότητας. Προσπαθούμε να επιτύχουμε κάποια πράγματα ε, στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, κάποια άλλα περιβαλλοντικά, κάποια άλλα θέματα εργασιακά. Και επίσης, δείχνει και το ζήτημα της δημοκρατίας. Όπως ξέρετε, οι εμπορικές μας συμφωνίες είναι κάτι το οποίο προωθούμε ως υποστηρικτικό ε, για μια συνεργασία σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο που να βασίζεται ε, σε κανόνες και να είναι προβλέψιμο και γενικότερα να δημοκρατικές συγκοινωνίες. Ένας άλλος τίτλος είναι η ευημερία και αποτελεί και συνέχεια. Είναι μια μόνιμη εποδός ε, στη συνεργασία μας με τη Λατινική Αμερική και στις διαπραγματεύσεις οι οποίες τρέχουν με τη Χιλή για παράδειγμα οι συμφωνίες εφαρμογής με την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό και το Μεξικό και έχουμε και την ολοκλήρωση ε, των ε, συμφωνιών με τη Μερκοσούρ. Από την ανακοίνωση θα δείτε ότι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή ήταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας Μερκοσούρ. Και ευτυχώς καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολιτικά συμπεράσματα στο διάστημα ανάμεσα στην έγκριση αυτής της ανακοίνωσης και τη σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, δεν θέλω να σας ε, κουράσω και να μακρηγορήσω. Όπως είπα προηγουμένως, το εμπόριο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική. Βασικά δύο στοιχεία ανακλώνται στην ανακοίνωση αυτή. Πρώτον, το εμπόριο, τα οικονομικά και οι αξίες και μετά το άλλο βασικό στοιχείο είναι η πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, το όραμα που έχουμε με τη Λατινική Αμερική. Να έχουμε μια εταιρική σχέση πολύ ευρύτερη από την αμυγός εμπορική. Σε αυτή την ανακοίνωση αυτό θέλησαμε να αναπτύξουμε και να παρουσιάσουμε Και όπως βλέπετε συμπεριλαμβάνουμε το εμπόριο σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κεφάλαια της ε, ανακοίνωσης. Το εμπόριο δεν είναι κάτι το αυθύπαρκτο, δεν είναι ότι έχουμε μια συμφωνία με ένα εμπορικό πυλώνα. Θέλουμε να πούμε ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, ενσωματωμένη σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής, γιατί είναι ξεκάθαρο για μας ότι όλο και περισσότερο θα έχουμε αιτήματα για συνοχή και συνέπεια και συνέχεια της εμπορικής πολιτικής με άλλες πολιτικές όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάπως διαφορετική τώρα η θεώρηση και το όραμα που έχουμε σε σύγκριση με προηγούμενες ανακοινώσεις που ήταν ξεκάθαρη και χωρισμένη οι ε, διάφοροι πυλώνες. Τώρα είναι πιο ενιαία αντιμετώπιση, γι' αυτό χρειάζεται ε, συνέπεια, συνέχεια και αλληλοϊποστήριξη των διαφόρων κλάδων της πολιτικής. Ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εδώ παρούσα, και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση, ΔΕΦΚΟ φυσικά, αλλά και άλλους, όπως είναι η Γενική Διεύθυνση MOVE, γιατί έχει σημασία, ας πούμε, ο κλάδος των αερομεταφορών ή τη Γενική Διεύθυνση Connect που ασχολείται με την ψηφιακή οικονομία κτλ. Έχουμε όμως εδώ μία γερή βάση για ε, τις μελλοντικές μας εμπορικές σχέσεις και σε ένα συνολικό πλαίσιο συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική, πάντα με συνοχή και συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κλάουντα Γκίντερ από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τμήμα σχέσεων με τη Λατινική Αμερική. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ήδη ανέφερε ο Ματίας, η ανακοίνωση αυτή ήταν μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, έτσι ώστε να φανεί μια κοινή προσέγγιση. Πολύ συχνά το ε, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι κάτι που να μην μας δίνει ένα ευρύτατο όραμα, διότι συλλέγονται σε ένα σύστημα όλα τα μέσα που διαθέτουμε και από την άλλη η κοινή ανακοίνωση είναι ένα από τα πιο πρόσφατα έγγραφα στρατηγικής που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο θεωρούμε ότι η έγκριση του εγγράφου αυτού έχει έρθει στην πλέον κατάλληλη στιγμή, διότι το προηγούμενο έγγραφο των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική έχει ήδη κλείσει 10 χρόνια ύπαρξης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Καραϊβική, έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος ε, σε θέματα ανάπτυξης. 50 ε, εκατομμύρια πολίτες έχουν βγει από τη φτώχεια και έχουν αλλάξει λοιπόν τα δεδομένα. Αυτό έδειξε ότι υπήρχε πλέον ανάγκη να ξεπεράσουμε την παραδοσιακή συνεργασία και να προσανατολιστούμε σε μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων. Ταυτόχρονα, πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα αναπτυξιακά και χρειάζονται τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη και τη δική μας ε, συνεργασία. Φυσικά, ε, είναι γνωστό ότι ορισμένες χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα περνάνε περίοδους μεγάλης κρίσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η στρατηγική χρειάζεται ευελιξία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ε, ανάγκες και στις συγκυρίες της εκάστοτε χώρας. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους ε, της ευελιξίας αυτής είναι η ποικιλομορφία. Από την άλλη, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αναφέρομαι στο ΣΕΛΑΚ, το οποίο στην ε, Βενεζουέλα χωρίστηκε, δεν ε, ήταν δυνατόν να βρεθεί μια κοινή θέση και δεν ε, είχε γίνει σύνοδος από το 2015 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΣΕΛΕΚ. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να βρεθεί ένας διαφορετικό τρόπος να γίνουν συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο χωρίς να οδηγηθεί σε αδιέξοδο η διαδικασία ολοκλήρωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους της ανακοίνωσης, Νομίζω πως καταρχάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαίο να επαναληφθεί η δέσμευσή της ε, για την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι κάτι που θεωρούσαμε δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι πάντα αναφερόμασταν σε κοινωνικούς δεσμούς, ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή αυτή. Όμως ε, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, δεν έχουν γίνει ε, αποστολές υψηλού επίπεδου και αυτό εξηγείται με το ότι στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κρίσεις που ε, χρήζουν προσοχής. Χρειάζεται όμως ε, να δείξουμε το παρόν στην περιοχή αυτή, να υποστηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την Κούβα και τέλος φυσικά να προσπαθήσουμε να μεσολαβήσουμε για να λυθούν τα προβλήματα στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακυβεύονται στην περιοχή αυτή. Για πολλές ε, χώρες της ε, Λατινικής Αμερικής η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος και συνολικά είναι ο τέταρτος σημαντικότερος παγκοσμίω. Πολλοί νέοι, 15 έως 25 ετών, τα επόμενα δέκα χρόνια θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις χώρες τους να πλουτίζουν μετά την αύξηση της ε, συνεργασίας. Έπειτα, οι σχέσεις με την Καραϊβική αντιμετωπίζουν διάφορες ε, προκλήσεις, ε, διότι μετά από την μεταναστευτική κρίση που προκλήθηκε από την κατάσταση στην Βενεζουέλα υπάρχει και το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, πολλές από αυτές τις χώρες ε, είναι δυνητικοί εταίροι. Μπορούν να ε, συμμεριστούν τις ε, ίδιες αξίες και να στηρίξουν τις ίδιες προσπάθειες. Αυτά φυσικά είναι πολύ γενικά, διότι οι θέσεις και οι κυβερνήσεις αλλάζουν, όμως πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα, διότι αναζητούμε εταίρους σε πολυμερή φόρα. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο να στείλουμε ένα μήνυμα και να προχωρήσουμε και ε, για χάρη του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Υπάρχουν ανταγωνιστές όπως η Κίνα οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια δυνατή βάση στην περιοχή, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και βλέπουμε ότι οι Κινέζοι δεν σταματούν εδώ, θα συνεχίσουν έτσι ώστε να αποκτήσουν το προβάδισμα. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί προσοχή σε αυτό, καθώς και στο ότι προσπαθούν να βελτιωθούν οι σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Μετά, η ανακοίνωση επίσης προσπάθησε να αντλήσει διδάγματα από τις ε, εμπειρίες του παρελθόντος και να ενημερώσει την, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο για την κατάσταση από το 2021 έως το 2027 θα δρομολογηθεί κατά πάσα πιθανότητα και το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Αυτά προς το παρόν. Συνοπτικά η κοινή ανακοίνωση προσβλέπει σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής τα επόμενα 10 χρόνια σε τομείς ε, τους οποίους θεωρούμε πολύ σημαντικούς. Και τέλος ο τρόπος που θα γίνει αυτή η συνεργασία με συγκεκριμένα ε, βήματα. Υπάρχει μία δομή πάνω στην οποία θα βασιστεί αυτή η συνεργασία. Ο Ματίας αναφέρθηκε στον κοβανά της ευημερία σε, ένα, μια διαδρομή προς ε, πιο φιλική σχετικά προς το περιβάλλον μέτρα, σε ενίσχυση του εμπορίου και φυσικά στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και στις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ένας άλλος πολύ σημαντικός ε, τομέας είναι η δημοκρατία, η οποία δεν είναι δεδομένη. Δεν νομίζω πως πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε κανένα σημείο του κόσμου, πόσο μάλλον στη Λατινική Αμερική, όπου ε, έχει αυξηθεί ο σκεπτικισμός των πολιτών απέναντι στην ε, δημοκρατία, στις ε, διαδικασίες όπως οι εκλογές κτλ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να στηρίξουμε την δημοκρατία στη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι ιστορικό μας καθήκον, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου χρειάζεται περισσότερο. Φυσικά έχουν ξεσπάσει διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς που υπονομεύουν τη δημοκρατία, γι' αυτό και θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά μας η καταπολέμηση της διαφθοράς. Και να μην ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προασπίσουμε σε όλες ε, τις ε, πτυχές, όχι μόνο τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και των ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα στις μεταξύ μας σχέσεις. Τέλος, άλλο σημαντικός τομέας, η ανθεκτικότητα. Είναι μια αφηρημένη έννοια κατά κάποιον τρόπο, όμως μας λέει πολλά. Ε, πρόκειται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, για την αύξηση της ασφάλειας των πολιτών, καταπολέμηση των ναρκωτικών και της διακίνησης. Γιατί όπως γνωρίζετε η Λατινική Αμερική είναι ε, από τις πιο προβληματικές ε, περιοχές στο τομέα αυτό, η οποία μαστίζεται και από φτώχεια. Και τέλος είναι η αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση ένας πολύ σημαντικός τομέας. Αναζητούμε εταίρους παγκοσμίω και η Λατινική ε, Αμερική είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτη αυτό. Αποτελεί υπολογίσιμη δύναμη σε όλα τα διεθνή φόρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί αυτή η ιδιότητα. Το έγγραφο λοιπόν, όπως ε, ήδη ανέφερα, εστιάζει τα ε, κοινά που έχουμε, ψηφιακή συνεργασία, ψηφιακή οικονομία, καινοτομία, εμπόριο, επενδύσεις, κοινέ αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα. Η περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου προκλήσεις. Χρειάζεται να προσαρμοστούν οι πολίτες στις ε, καταστροφές που είτε είναι φυσικές είτε έχουν προκληθεί από τον άνθρωπο και να σας θυμίσω ότι την πιο πρόσφατη από αυτή, τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Όπως ακούστηκε δε, και πριν, δεν υπάρχει πλέον το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΛΑΚ, Υπάρχει όμως μια ευελιξία που αναφέρεται στην ανακοίνωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τις χώρες αυτές οι οποίες το επιθυμούν, οι οποίες επιθυμούν μια στενότερη συνεργασία, για παράδειγμα, όπως ε, για παράδειγμα με τη Συμμαχία για τον Ειρηνικό που, με την οποία πρόσφατα υπογράψαμε με κοινή δήλωση. Και για να ολοκληρώσω, η κοινή δήλωση δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μάλλον μια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και να εντοπίσουμε τις επόμενες κινήσεις για τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη. Η κυρία Ραφαέλα είναι πρώτη. Ευχαριστώ πολύ για την ανακοίνωση αυτή και την παρουσίαση. Εκτιμώ ε, όλα αυτά. Τις ε, τελευταίες εβδομάδες ε, επισκέφτηκα τις Ολλανδικές υπερπόντιες περιοχές, την Αρούμπα, το Κουρασάο και εκτιμώ ιδιαίτερα την έκκληση για την εξωτερική διάσταση των ε, πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναρωτιέμαι γιατί η πρόσφατη κατάσταση των υπερπόντιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνηση. Και για να είμαι ειλικρινής, ε, έχω λίγο την εντύπωση ότι οι υπερπόντιες περιοχές είναι κάπως ξεχασμένες στην ανακοινωσή σας και θεωρώ εν γέννη όταν συζητούμε το θέμα αυτό ε, τις ξεχνάμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και την άποψή σας επ' αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μακουλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχω? Όσο θέλετε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση ε, του εγγράφου και για την ε, εκπόνησή του και την όλη δουλειά που κάνετε γενικότερα. Θα ήθελα να κάνω διάφορες ερωτήσεις ε, για διαφορετικά ζητήματα. Καταρχάς, όσον αφορά την Κεντρική Αμερική, από το 2015 ισχύει η συμφωνία, αλλά έχουμε καταφέρει μόνο να εφαρμόσουμε το εμπορικό σκέλος, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει τα κοινοβίλια τους για να ε, ε, ε, τεθεί σε ισχύ το θέμα σύνδεσης και συνεργασίας. Τι μπορεί να γίνει ώστε να μην πλήξει τους πολίτες της Κεντρικής Αμερικής η κατάσταση. Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε με τις μελλοντικέ συμφωνίες σύνδεσης. Πώς μπορούμε να, δούμε, να δώσουμε όθηση ώστε να κυρωθούν οι συμβάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και έχουν ακυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την Ικαράγουα, φέτος με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στην Ικαράγουα, όπου ζητούσαμε την ενεργοποίηση της δημοκρατικής ρήτρας της συμφωνίας και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση στην οποία ο εθνικός διάλογος ε, δεν θα οδηγούσε σε αποτελέσματα ε, τα οποία περιμέναμε. Η κατάσταση στην Ικαράγουα έξι μήνες μετά δυστυχώς δεν έχει αλλάξει και θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το σχέδιο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε οι πολίτες της Νικαράγουας ε, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη δημοκρατία, τις ε, ε, ελευθερίες τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ακόμα έχουμε και πολιτικούς αντιφρονούντες στις φυλακές την Κούβα. Όταν ε, τελείωσε το ε, μορατόριο του νόμου Χέμς Μπάρτερ ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν κάποιοι περιουσίες οι οποίες τους είχαν στερηθεί εδώ και 70 χρόνια. Ε, συζητούνται πιθανές κυρώσεις ώστε η προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να ε, τύχει υπεράσπιση. και ορισμένα ε, εξετάθηκε και το ενδεχόμενο ε, να υπάρχει μπλόκο. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την επιπλέον επίθεση από πλευράς του Τραμπ που είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Για το Μερκοσούρ θα ήθελα να ξέρω πότε θα είναι διαθέσιμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κείμενο της συμφωνίας, πότε θα δημοσιευθεί και η αξιολόγηση επιπτώσεων, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας εμείς οι Ευρωβουλευτές και κυρίως το τι κάνει η Επιτροπή μας. Τώρα, στην Κολομβία μόλις μάθαμε ότι οι ΦΑΡΚ ξαναπήραν τα όπλα και θα ήθελα να ξέρω ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Κολομβία για την εφαρμογή, όλη τη διαδικασία ε, συνεργασίας και όλα τα όσα συμφωνήσαμε μαζί τους για, τη συμφωνία των, ε, για την εφαρμογή των συμφωνιών της ειρήνης. Για το Μεξικό. Πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί ο κατάλογος ε, για τις δεσμεύσεις, για τα θέματα των ε, δημοσίων συμβάσεων και να ληφθούν υπόψη όσα έχουν συμφωνηθεί και να μπορέσουμε ε, να δούμε και τι έγινε στο Μεξικό για το Κοινοβούλιο. Ε, για τη Χιλή, τι γίνεται με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τη Χιλή, πώς έχουν συγκεκριμένα τα θέματα Ε, ισότητα των φύλων και τι μπορούμε να κάνουμε για τα περισσότερα θέματα της Λατινικής Αμερικής ε, για να βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες για να μπορέσουν ε, να εκμεταλλευτούν αυτές τις συμφωνίες εμπορίου. Ευχαριστώ και... Τώρα, η κυρία Βεντρέν, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύτερο όραμα δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ούτε από τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε από την ανάπτυξη το εμπόριο. Και πολύ σωστά είπατε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περιοχή αυτή για εμάς και θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη σχέση μας και θα είναι και υποστηρικτική στην πολυμερή συνεργασία. Ε, συνεχίζω από αυτά που είπε η συνάδελφος Ραφαέλα για να αναφερθώ στο μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες που την 1η Πρώτου του 2020 εκπνέει. Πέρα από τον ΠΟΕ που υπάρχει ένας μηχανισμός, θα ήθελα να μάθω τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει είτε την ανανέωση αυτού του μηχανισμού είτε ένα νέο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπριγμό. Ε, Ευχαριστώ. Ε, κυρία μου, για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τα θετικά, στα οποία δεν θα επανέλθω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά στην ανακοίνωση αυτή υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία που θα πρέπει να αναδειχθούν, αλλά και ερωτηματικά. Υπάρχει ένα θέμα που κάπως γρήγορα το διεκπεραιώνει ε, η ανακοίνωση, που είναι ε, η χρηστή διαχείριση των φορολογικών. Από το Μάρτιο ε, το ΕΚΟΦΗΝ του 2019 ε, η μαύρη λίστα πέρασε από τις 5 χώρες στις 15 και από τις 15 αυτές, 5 είναι χώρες Καραϊβικής. Η μαύρη λίστα του Συμβουλίου, του ΕΚΟΦΗΝ, ε, για τα φορολογικά, τους φορολογικούς παραδείσους. Επίσης υπάρχουν νέες συμφωνίες που αυτό το καιρό διαπραγματευόμαστε για τις αερομεταφορές, για να ανοίξουν νέες οικονομικές δυνατότητες και νέες αγορές και δεδομένων και των συζητήσεων που είχαμε σήμερα το πρωί, θα ήθελα να επιμείνω στη συνοχή και την συνέπεια των πολιτικών μας ε, και πώς αυτές συνάδουν με ε, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τους στόχους Συμφωνίας των Παρισίων. Γιατί βλέπω λίγο κάποια αντιφατικά ε, εδώ να ισχύουν σε σχέση με τις δηλώσεις ο τίτλος επίσης ε, της ανακοίνωσης μου κάνει εντύπωση. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα κοινό μέλλον. Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνέπεια και συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές μας. Και κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε ε, αυτή την περιφέρεια ως ένα τεράστιο χώρο ε, πρόσβασης για φυσικούς πόρους για μας και μια τεράστια αγορά. Θα πρέπει να είμαστε πιο δεσμευτική ε, ως προς την ε, υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά όταν ψάχνουμε νέες αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά μου, λέει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να πω το εξής. Νομίζω αναφερθήκατε έτσι επιγραμματικά κάπως στην Κίνα σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, είναι το μεγάλο ταμπού η Κίνα που δεν αναφέρει κανείς. Έχουμε πολλά έργα υποδομών που κατασκευάζουν στη Λατινική Αμερική ε, κινέζικες εταιρείες. Έχουμε δει επίσης και πάρα πολλά κινέζικα προϊόντα να κυκλοφορούν εκεί, στη Λατινική Αμερική. Και οι κινέζικες εταιρείες ε, ε, ε, συμμετέχουν στην εξόριξη λιθίου στη Χιλή. Το λίθιο είναι απαραίτητο για τις μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τα λοιπά. Συμφωνώ απολύτως με την ανακοίνωση ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο και να προσέξουμε περισσότερο αυτή την περιοχή του κόσμου γιατί ήταν πάνω κάτω δεδομένο το θεωρούσαμε ότι θα έχουμε στενέ σχέσει. Βεβαίω έχουμε ισχυρού δεσμού, ε, ιστορικούς και πολιτισμικού με την περιφέρεια αυτή. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό από πλευρά τη Κίνα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα μα βοηθήσουν να έχουμε καλύτερου εμπορικού δεσμού με την Λατινική Αμερική. έτσι ώστε να έχουμε μια εταιρική σχέση που να βασίζεται σε κοινέ αξίες και αυτά να υπερτερούν σε σχέση με κάποια οικονομικά συμφέροντα από πλευρά της Κίνας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Ο Ματίας. Ε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην ε, κυρία Ροντρίγκη Πινιέρο, η οποία ρώτησε για το χρόνο που έχουμε. Ήταν πολλές ε, και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κάποιες έμεσες, κάποιες και άμεσες. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όμως με τη σειρά που έγιναν. Σε ό,τι αφορά τις ε, υπερπόντιες ε, περιοχές και δάφη δεν θα έλεγα πως είναι ξεχασμένα εδάφη, είναι κομμάτι αναπόσπαστο της συνολικής μας στρατηγικής για την περιοχή και να είστε σίγουροι ότι στις εμπορικές μας συμφωνίες φροντίζουμε έτσι ώστε προϊόντα όπως οι μπανάνες ή η ζάχαρη που είναι πολύ σημαντικά προϊόντα για τις περιοχές αυτές δεν είναι αντικείμενο πλήρους απελευθέρωσης, αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί με το άνοιγμα της αγοράς. Ε, πολλές φορές με έλεγχο ή με μερική απελευθέρωση, όπως ε, για παράδειγμα έγινε με τη μπανάνα. Εκεί οι εμπορικές σχέσεις με την ε, Λατινική Αμερική θα παραμείνουν σταθερές και από το τέλος του έτους θα υπάρχει ένας μόνιμος εδασμός 75 ευρώ ανατόνο για την εισαγωγή μπανάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε λοιπόν πρόθεση να προχωρήσουμε σε περαιτέρω απελευθέρωση στο τομέα αυτό. Ακόμα και αν ο μηχανισμός σταθερότητας ε, της τιμής της μπανάνας θα λήξει στο τέλος του 2019. Και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το ότι δεν θα πλημμυρίσει η αγορά με μπανάνες. Βλέπουμε τις εμπορικές τάσεις των τελευταίων ετών, τις παρακολουθούμε προσεκτικά και παρατηρήσαμε ότι η εισαγωγή μπανάνας δεν έχει αυξηθεί, ούτε έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα που θα πυροδοτούσαν την ε, χρήση του μηχανισμού σταθεροποίησης και την πιθανή επιστροφή σε υψηλότερους δασμούς. Όμως να είστε σίγουροι πως παραμένουμε σε επαγρύπνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και είμαστε έτοιμοι να θέσουμε σε ισχύ τις διαφορές ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία επικύρωσης στην Ευρώπη. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να συνεχίσουμε την πίεση στα κρατη έτσι ώστε να προχωρήσουν διότι η συμφωνία αυτή θα αυξήσει την αξιοπιστία μας στην, ε, στον υπόλοιπο κόσμο, στην Λατινική ε, Αμερική. Δεν πρέπει να χρειάζονται 7-10 χρόνια μέχρι την επικύρωση μιας συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε Πώ θα επιταχύνουμε τη διαδικασία. Είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσουμε επίσης τους εταίρους μας ε, το πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία όταν ε, μα παίρνει πάνω από 10 χρόνια για να την ολοκληρώσουμε. Επόμενη ερώτηση ήταν πότε θα είναι έτοιμο προς ε, αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κείμενο για τη Συμφωνία Mercosur. Πρώτα χρειάζεται να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα των συζητήσεων. Υπάρχουν κάποια προσχέδια που έχουμε αυτή τη στιγμή, όμως να είστε σίγουροι ότι θα διατηρήσουμε το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θα δημοσιεύσουμε το κείμενο το συντομότερο, μόλις το έχουμε και εμείς. Η διαδικασία λοιπόν της ενομικής αναθεώρησης έχει μόλις ξεκινήσει. Αυτό όπως γνωρίζετε θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά αναμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή κάποια στιγμή στο πρώτο μισό του 2020. Κατόπιν με το που γίνουν οι μεταφράσεις θα σας ε, παρουσιάσουμε την επίσημη πρόταση. Μετά. Μεξικό. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με το Μεξικό για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο για, τις, ε, για τα διάφορα ομόσπονδα κράτη του Μεξικού. Φυσικά και εμείς επιθυμούμε η συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας ε, δώσουμε την τελική πρόταση νομίζω πως είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Είναι σίγουρα για μας προτεραιότητα να φτάσει το γρηγορότερο δυνατόν στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να επικυρωθεί και να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο. Ε, με την Χιλίνο τώρα, νομίζω πως οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Έχουμε έναν εταίρο ο οποίος έχει δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή του. Τον Ιούλιο λάβαμε την έκθεση, έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Ο των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει μάλλον τον Νοέμβριο. Η πρόοδος είναι αρκετά σημαντική. Χτίζουμε πάνω σε αυτά που ήδη έχουμε επιτύχει από τον Ιούλιο και έπειτα, αλλά αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ε, δύσκολα θέματα, όπως για παράδειγμα το επενδυτικό δικαστήριο, οι γεωγραφικές ενδείξεις ε, και άλλα. Σε ό,τι αφορά τώρα το εμπορικό θεματολόγιο και εδώ έχει σημειωθεί πρόοδος παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μας ακόμα. Είμαι όμως αισιόδοξο ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, θα υπάρχουν δεσμεύσεις και ένας μηχανισμός επιβολής και αυτό μάλιστα είναι κάτι που βλέπουμε και από την πλευρά της Εχιλής υπάρχει έντονη δέσμευση και προθυμία. Με την Κίνα τώρα νομίζω πως έχετε απόλυτο δίκιο που αναφερθήκατε στο θέμα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με την Λατινική Αμερική απέναντι στην Κίνα. Νομίζω πως ε, το πλαίσιο που έχουμε είναι αρκετά καλό και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όταν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Μερκοσούρ. Αυτό που απομένει είναι να δούμε και τα υπόλοιπα μέσα που διαθέτουμε, για παράδειγμα τις δυνατότητε δανειοδότησης, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτήν την καλή σχέση με τη Λατινική Αμερική. Και είναι ξεκάθαρο πως ε, αν η μία πλευρά αφήσει κενά και αν υπάρχουν αυτά τα κενά κάποιες άλλες χώρες θα σπεύσουν να τα καλύψουν. Γι' αυτό χρειάζεται δουλειά ακόμα, διότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Αν δεν είναι η Κίνα αυτή, θα είναι κάποιος άλλος. Νομίζω πως έχω απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις. Α, ίσως να απαντήσω σε σας Αγαπητέ συνάδελφε, ναι, συμμερίζομαι και εγώ την ανησυχία σας. Έχουμε ένα αρκετά κανό πλωστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τις ε, εξωτερικές προκλήσεις, όπως τώρα με τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν θα διστάσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Για παράδειγμα, ε, το μπλοκάρισμα που αναφέρεται. Ματίας, μου έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι το λόγο. Η κυρία Ραφαήλα και η Έμα. Ναι, ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ ρωτούσα για την ευρύτερη σημασία των υπερπόντιων περιοχών και όχι μόνο κάποια μεμονωμένα προϊόντα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ε, τι όραμα έχετε εσείς για το πώς μπορούν να συμμετέχουν και οι υπερπόντιες περιοχές, διότι αναφερόμαστε στο εμπόριο και το μελλοντικό, το κοινό μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να έχω ένα πιο ρητό όραμα για το πώς μπορούν να συμμετέχουν και οι υπερπόντιες περιοχές ε, σε θέματα εμπορίου. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία δεν απαντήσατε. Ευχαριστώ για όσα μου απαντήσατε, αλλά ε, για την Ικαράγουα. Δεν ξέρω ακριβώς ε, τι δυνατότητα υπάρχει να ενεργοποιηθεί η δημοκρατική ρήτρα και να ε, υπάρξουν κυρώσεις εάν δεν προχωρήσουν τα θέματα ε, με το Εθνικό Συμβούλιο. Ε, για την Κούβα επίσης δεν μου είπατε για το τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση του νόμου Χέμου Μπάρτον από τις Ηνωμένε Πολιτείε και επίσης δεν μου είπατε τίποτα για την κατάσταση στην Κολομβία και πώς μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή εν ώψη κυρίως και της ενεργοποίησης πλέον των ΦΑΡΚ και της επιστροφής στα όπλα. Ματίας, ναι, ευχαριστώ. Το πρώτο είναι θέμα της συνολικής ε, αναστολής ε, της συμφωνίας που είναι πολιτικό ζήτημα. Και νομίζω ότι έγιναν συζητήσεις ε, στο κόλακ για το θέμα αυτό. Με την άδειά σας λοιπόν θα απαντήσει η Για την Κούβα το σημείωσα, νομίζω ότι απάντησα, αλλά σημείωσα την άποψή σας επί του θέματος. Και για την Κολομβία, αν κατάλαβα καλά το τελευταίο σημείο ήταν για την Κολομβία. Και εδώ θεωρώ ότι είναι ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς από πλευράς εμπορίου είναι ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική σχέση που έχουμε και αυτό περιλαμβάνει και τη Συμφωνία Εμπορίου για να είναι πιο δελεαστικό για τους Κολομβιανούς και την Κολομβία να σταματήσει να παράγει ε, ναρκωτικά και να φυτέψει και να καλλιεργήσει και να εξάγει άλλα προϊόντα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Το, ε, δεν ξέρω αν η Κλάουντια θα έχει κάτι να προσθέσει. Ανησυχούμε ιδιαίτερα από τον αρνητικό ε, αντίκτυπο στο εμπόριο και το επενδυτικό κλίμα. Φυσικά και μας ενδιαφέρει, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προωθήσουμε την εμπορική συμφωνία ώστε να είναι δελεαστική για τα θέματα αυτά. Τώρα, για τις υπερπόντιες περιοχές, τις εξόχως απομακρυσμένες. Δεν είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, υπάρχει πύρης πρόσβαση στις αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις περιοχές. Προστατεύουμε ευαίσθητα προϊόντα από τις περιοχές αυτές ε, στις εμπορικές μας συμφωνίες με άλλους. Σημειώνω την ανησυχία σας, θα την παραπέμψω στους αρμοδίους και πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε και διμερώς ε, και με άλλους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που ίσως ε, να γνωρίζουν πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα για το θέμα. Ευχαριστώ. Η Κλάουδια. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, δεν μπορέσω να τις απαντήσω όλες, 100% ικανοποιητικά για σας. Μόλις ε, επέστρεψα από μια αντιπροσωπεία και είναι η δεύτερη μέρα μου σήμερα εδώ. Δεν σημαίνει όμως ε, ότι μου ήταν άγνωστα αυτά τα θέματα. Στη Βραζιλία υπηρετούσα μέχρι τον περασμένο μήνα και τώρα ε, σήμερα ήδη ανέλαβε ο νέος πρέσβης στη Βραζιλία. Ο Ματίας επίσης απάντησε και για άλλες χώρες και για τη Βραζιλία. πρέπει να δούμε τι προγραμματίζουν και τι θα κάνουν μαζί μας και κατά πόσο είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Βεβαίως μας ανησυχεί πολύ η κατάσταση και δραστηριοποιούμεθα. Για την Νικαράγουα φοβάμαι ότι δεν έχω τις τελευταίες εξελίξεις. Φυσικά μέσω του διαλόγου και των ε, ελεύθερων ε, δημοκρατικών εκλογών λύνονται τα θέματα, αλλά εξετάζουμε και όλα τα ενδεχόμενα, μπορεί και κυρώσεις να χρειαστούν. Θα επανέλθω. Ε, εάν υπάρχει τίποτα νεότερα να σας ενημερώσω. Πάντως αυτή είναι η γενική μας θέση για την κρίση στην Ικαράγουα Και δεν υπάρχει πρόοδος στο παρά. Για την Κολομβία μπορεί να είδατε ε, ότι υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως υποστήριξε την ειρηνευτική διαδικασία και θα εξακολουθήσει να το πράττει. Η απόφαση απόσυρσης από τη διαδικασία αφορά μόνο λίγα μέλη των ΦΑΡΚΑ, και σε ό,τι μας αφορά αυτή τη στιγμή παραμένει ενισχύει η νευτική διαδικασία και εξακολουθούμε να την υποστηρίζουμε, αλλά φυσικά παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την ε, κατάσταση και κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Για την Κίνα βεβαίως πραγματικά έχετε δίκιο, είναι ένα θέμα ταμπού που όλοι το ξέρουν και κανείς δεν το αναφέρει. Καλό είναι όμως να ολοκληρωθεί η συμφωνία Μερκοσούρ, γιατί αυτό θα μας ισχυροποιήσει και θα βοηθήσει και θα κάπως θα είναι ένα ε, αντιπαλωδέος στις ε, κινέζικες επενδύσεις. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δείχνουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, τις εργασιακές ε, νομοθεσίες και υπάρχει και η κοινωνική εταιρική ευθύνη παράδειγμα που δείχνει ότι έχουμε και ποιοτική διαφορά. Ε, ε, δηλαδή οι ευρωπαϊκές επενδύσεις και οι κινητικές επενδύσεις δεν είναι το ίδιο. Και αυτό το μήνυμα το κατανοούν και οι εταίροι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ λοιπόν η σύντομη συζήτηση για αυτό το θέμα που δεν είναι η τελευταία φορά που θα τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. No, unfortunately we can't... Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε το λόγο. Αλλιώς θα ήθελα να πάρουν όλοι το λόγο, καταλαβαίνετε. Την άλλη φορά θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποιες χώρες και θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Στις 15. Πάντα το Κοινοβούλιο ε, ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει με τους κανόνες ε, για την ονομασία προέλευσης, ε, για τις προέλευση των εμπορευμάτων. Um, if anybody wants to leave the room, please. Παρακαλώ ποιος θέλει να φύγει ήσυχα. So, the rules of... Τι είναι κανόνες προέλευσης. Καμιά φορά εφιάλτης. Γιατί αλλάζουν άλλαξαν το 2017, όχι πάρα πολύ διαφανώς πάντα. Το 2017 λοιπόν κάναμε μια κρόση εδώ στο Κοινοβουλίο για να ρίξουμε λίγο φως σε αυτό το σκοτάδι. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει και πώς έχουν οι εξελίξεις ε, σχετικά ε, με αυτό το θέμα τα τελευταία έτη και τι γίνεται με την εφαρμογή. And of course, Και πώς θα αλλάξουν στο μέλλον. Υπάρχουν κάποια α, είδη πάρα πολύ ε, αμφιλεγόμενα, ε, όπως ε, στο Μερκοσούρ το θέμα των αυτοκινήτων, ξέρω. Θα δώσω το λόγο στην αρμόδια ε, διεύθυνση και στο αρμόδιο τμήμα στον Ιγνάσιο και δεν θα σας πω το επίθετο γιατί δεν το βγάζω. Ε, θα αφήσουμε Ιγνάτιο. Είναι περίπλοκο βάσκικο όνομα το επίθετό μου. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία ε, να παρουσιάσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ε, κανόνες προέλευση ήταν δικό σας αίτημα και ερχόμαστε να απαντήσουμε σε αυτό. Για να εξηγήσουμε την πρακτική και πώς ε, άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία θα σας παρουσιάσω στην αρχή του εγγράφου και μετά με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Οι προτιμησιακοί κανόνες προέλευσης είναι ένα απαραίτητο συστατικό σε οποιαδήποτε συμφωνία προτιμησιακού χαρακτήρα. Αν δίνουμε ευνοϊκές δασμολογικές ρυθμίσεις σε μία χώρα ή σε μία περιφέρεια, θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε και να εξακριβώνουμε αν όντως προέρχονται από τις χώρες αυτές ε, ή από αλλού τα προϊόντα. Και θα πρέπει πάντα να βεβαιωνόμαστε ότι η επεξεργασία τους, η κατεργασία τους, η παραγωγή τους έχει γίνει στις χώρες με τις οποίες έχουμε προτιμησιακό καθεστώς. Συνοψίζοντας, τι κάνουμε συνήθως για τους κανόνες προέλευσης. Καθορίζουμε ένα κατόφλι οικονομικής δραστηριότητας και θα επανέλθω σε αυτό τι σημαίνει ε, κατά την παραγωγή ενός προϊόντος, κατά την κατασκευή του και βάζουμε κανόνες για το πώς ε, ελέγχεται αυτή η δραστηριότητα. Να αρχίσω από το επίπεδο Πώς ορίζεται αυτό το κατόφλι ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα για την παραγωγή ενός προϊόντος σε μια χώρα όπου έχουμε προτιμησιακή συμφωνία. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και στην παγκόσμια λυσίδα παραγωγής. Ας πούμε, ε, όταν έχεις ένα μηχάνημα μπορεί τα ε, διάφορα ανταλλακτικά του να παράγονται σε διαφορετικές χώρες ή τα εξαρτήματα. Ε, σήμερα ένα περίπλοκο μηχάνημα δεν παράγεται κατά 100% ε, στην ίδια χώρα. Υπάρχουν ε, εξαρτήματα από άλλες χώρες. Αλλά όταν έχουμε προτιμησιακή συμφωνία με μία χώρα, αυτό αφορά τη συγκεκριμένη χώρα και μόνο και όχι την υπόλοιπη φίλιο και δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε και να επιτρέπουμε να θεωρείται προτιμησιακή σχέση όταν παράγεται το προϊόν κατά 0,001% εκεί. Γιατί θα μπορεί οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου να περνάει τα προϊόντα της από αυτή τη χώρα, να βάζουν τη τελευταία στρώση ε, βαφής και να το πουλάνε σαν προϊόν που έχει παραχθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Και να αποφύγουμε λοιπόν αυτές τις παρακάμψεις και τα τρίγωνα. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δημιουργήσαμε το 2011 όταν μεταρρυθμίστηκε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και αυτό το χρησιμοποίησαμε ως αφετηρία ε, στη διαπραγμάτευση των διαφόρων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από συμφωνία σε συμφωνία ε, ελευθέρου εμπορίου, γιατί κάθε φορά θα πρέπει να προσαρμόζουμε τη θέση μας και την τακτική μας απέναντι στους εταίρους της εκάστοτε χώρες και τελικά να αισθανόμαστε άνετα και οι δύο. Δεν είναι ε, καρμπών η ε, συμφωνία αυτή, η πλατφόρμα σε όλες τις χώρες, αλλά μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα γενικό κοινό πλαίσιο. Αυτό ήταν πραγματικά εξέλιξη. σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν το 2011. Δηλαδή τώρα πλέον είμαστε πιο ευέλικτοι από ό,τι στο παρελθόν και επιτρέπουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερα εξαρτήματα ε, για την παραγωγή ενός μηχανήματος, ας πούμε. Ένα μηχάνημα πριν το 2011 επιτρέπαμε μόνο 25 με 40% ε, των εξαρτημάτων να παράγεται από άλλη χώρα για να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παραχθεί, ότι έχει κατασκευαστεί η μηχανή, ξέρω εγώ, στην Κολομβία ή σε οποιαδήποτε χώρα. Είναι τυχαίο το παράδειγμα. Από το 2011 και μετά έχουμε φτάσει στο 50%. Δηλαδή ε, ε, επιτρέπουμε τα μισά εξαρτήματα και ανταλλακτικά να προέρχονται από άλλη χώρα και επίσης έχουμε βάλει και εναλλακτικές λύσεις ευέλικτες, ας πούμε, για ένα μηχάνημα. Έχουμε είτε το 50% είτε εάν έχει ε, υποστεί μια επεξεργασία ε, στη φάση παραγωγής, να μπορεί να αλλάζει το φορολογικό, το δασμολογικό μάλλον ε, κλιμάκιο. Στο παρελθόν ήταν πιο αυστηροί οι κανόνε, τώρα είναι πιο ευέλικτοι και υπάρχει και εναλλακτική πρόταση. Είναι πιο εύκολο δηλαδή το σύστημα. Για την αναπτυξιακή βοήθεια, για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, επιτρέπουμε μέχρι και 70% γιατί καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητές τους και είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι. Αυτό το αναγνώρισε και η ομάδα των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών στον ΠΟΕ και το έχει υιοθετήσει ως δικό του ε, μοντέλο. Ε, είδα πριν από λίγους μήνες ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο επενεί τους κανόνες της Ένωσης, ιδιαίτερα το 70% και ζητεί από τα μέλη τους να χρησιμοποιούν τους δικούς μας κανόνες, τα μέλη του ΠΟΕ, για τις προτιμησιακές ε, συμφωνίες. Από το 11 και μετά λοιπόν έχουμε γίνει πιο ευέλικτοι ως προς την ουσία και επίσης και ως προς τον έλεγχο πώς αποδεικνύεται αυτό και πώς επαληθεύεται η προέλευση δηλαδή. Στο παρελθόν η απόδειξη βασιζόταν είτε σε κρατικά πιστοποιητικά είτε σε δήλωση των εξαγωγέων. Σήμερα έχουμε περάσει τη δήλωση των εξαγωγέων, με φορά και στην δήλωση των εισαγωγέων. Αν θεωρεί ο εισαγωγέας ότι έχει αρκετή προφόρηση για να πιστοποιήσει ότι έχει παραχθεί κάπου το προϊόν, ταλώς. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει από τα κρατικά πιστοποιητικά και τη δήλωση του εξαγωγέα και έχουμε περάσει τη δήλωση του εξαγωγέα, ακόμα και δήλωση του εισαγωγέα. Πιο ευέλικτη ακόμα μορφή απόδειξης της ε, προέλευσης. Επίσης, επαληθεύουμε με διαφορετικό τρόπο για το ποιος αποφασίζει τελικά εάν το προϊόν την χάνει προτιμησιακής καταγωγής ή προέλευσης. Στην αρχή τον τελικό λόγο είχε η χώρα εξαγωγική. Τώρα, επειδή αυτό το επέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο, έχουμε αλλάξει. Το γεγονό ότι είχε τον τελευταίο λόγο εξαγωγική χώρα, αυτό δημιουργούσε κάποια προβλήματα και δυσκολίε. Ήταν δύσκολο για μας να ζητάμε από τους εισαγωγούς μας δασμούς και να τους συλλέγουμε αν θεωρούσαμε ότι ήταν λανθασμένη αυτή η δήλωση. Δηλαδή, εισάγουμε ένα προϊόν από μια τρίτη χώρα. Έχουμε ε, βάσιμες αμφιβολίες κατά πόσο έχει παραχθεί το προϊόν αυτό στη χώρα αυτή. Ζητούσαμε από μια κρατική αρχή ε, να αποφανθεί, αποφαινόταν και μας δέσμευε αυτό. Αυτό άλλαξε. Τώρα ε, οι τελωνιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποφαίνονται, έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε και τους δασμούς, τους διαφεύγοντες και τους ε, φόρους σε αντίθετη περίπτωση. Και πέρυσι περίπου κάναμε μια μελέτη μεταξύ των επιχειρήσεων για τους κανόνες προέλευσης και καταγωγής, τι έχουν να πούνε, να επικρίνουν, ποια είναι η ικανοποίησή τους. Και πρέπει να πω ότι ε, πολλές από τις εταιρείες που απάντησαν, που ήταν πάνω από χίλιες, φαίνεται να συμμορφώνονται. Μόνο το 13% είπαν ότι δεν μπόρεσαν να συμμορφωθούν ε, με τους νέους αυτούς κανόνες. Αλλά ζητούσαν και περισσότερη πληροφόρηση. Το 67% ας πούμε των απαντών τον ζητούσαν περισσότερη πληροφόρηση για την πρόσβαση στην αγορά. και ήθελαν περισσότερες προφορίες σε περισσότερες επίσημες γλώσσες ε, της Ένωσης, αλλά και σε πιο ευανάγνωστη μορφή, γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και τεχνική και ο κόσμος δεν την καταλαβαίνει πάντα. Αυτή την ιδιόλεκτο που έχουμε μια, μια μικρή εταιρεία, μια μικρομεσαία κανονική εταιρεία που δεν είναι εξοικειωμένη με αυτή τη γλώσσα δεν μπορεί πάντα να καταλάβει τι λέμε. Και το θέμα είναι όχι μόνο το καταλαβαίνουν, αλλά να εφαρμόζουν τους κανόνες και να υποφελούνται. Αυτά και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Thanks a lot. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον συνάδελφο από εσάς. Αν νομίζετε πως τα έχετε καταλάβει όλα, θα σας βάλω διαγώνισμα. Ωραία λοιπόν, φαίνεται πως όλοι είναι ενήμεροι για την κατάσταση. Ίσως από μένα κάποιες ερωτήσεις. Είχαμε συζητήσει και παλαιότερα τους ε, κανόνες προέλευσης σε σχέση με την Ιορδανία και την ε, ένταξη των προσφύγων στην ε, διαδικασία παραγωγής, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα με τις υπόλοιπες. Εσείς τι άποψη έχετε, ποια είναι η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ε, κανόνες προέλευσης και για την ε, προτιμησιακή χορηγησή τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα των προσφύγων. Έπειτα, δεδομένων των αυξανόμενων παγκόσμιων ε, αλυσίδων αξίας, όπως για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο που η αλυσίδα αξία του είναι χιλιάδες χιλιόμετρα και διέρχεται πολλά σύνορα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει δυνατότητα να δούμε το αν ε, ένα τέτοιο προϊόν είναι φυκτό να παράγεται σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την Ιορδανία και την ε, κατάσταση με τους πρόσφυγες, ε, νομίζω πως καταρχάς η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική. Έχουμε γνώση της ε, νομοθεσίας. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως βελτίωση. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη θέση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε στάδιο εξέτασης. Τώρα, μετά, ε, για το παράδειγμα που δώσατε με τα κινητά τηλέφωνα, νομίζω το παράδειγμά σας ήταν ιδανικό. Είπα στην αρχή ότι οι κανόνες προέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντικοί, μάλλον αναγκαίοι. Με την περίπτωση των τηλεφώνων ήμασταν αρκετά τυχεροί, διότι εξαιτίας της ε, συμφωνίας για τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις προτιμήσεις. Δεν επιβάλλουμε λοιπόν δασμούς ανεξαρτήτως προέλευσης στα κινητά τηλέφωνα. Βέβαια, ως μηχάνημα έχει νόημα η ερώτησή σας. Υπάρχουν πολλά εξαρτήματα, πολλά κομμάτια μέσα σε ένα μηχάνημα ε, και μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εξαρτημάτων μηχανών. Όταν λοιπόν υπάρχουν διάφορα επίπεδα προμηθευτών, η κατάσταση περιπλέκεται. Όταν πας από προμηθευτή σε προμηθευτή, γίνεται πιο δύσκολη η κατάσταση για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος να παράσχει τις ε, δηλώσεις προέλευσης από όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που αποτελούν ένα μηχάνημα για να διαπιστωθεί η προσθέμενη αξία του προϊόντος. Αλλά υπάρχει και ένας εναλλακτικό κανόνας. Αλλάζει δηλαδή η επικεφαλίδα, αλλάζει η κατηγορία του δασμού. Και λέμε ότι δεν γνωρίζουμε μένα από πού προέρχονται όλα τα εξαρτήματα, αλλά υπάρχουν αρκετά, αρκετά που υπάγονται στην κατηγορία τάδε, ας πούμε. Αν συνδυαστούν όλα αυτά τα εξαρτήματα και το αποτέλεσμα θα ε, υπάγεται σε άλλη κατηγορία, τότε ενδεχομένως να υπάρχει ευρωπαϊκή προέλευση όταν η τελική συναρμολόγηση έχει γίνει στην Ευρώπη. Βέβαια, όπως σας είπα, το η κατάσταση περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο και όσο μεγαλύτερος ο κατακαιρματισμός τόσο περισσότερο κατακαιρματίζεται και η λυσίδα αξίας. Παρομοίως και με μία εταιρεία, όταν ας πούμε κάποιος από τους εταίρους μας μας ζητά να διαπιστώσουμε εάν αυτά που δηλώνει μια εταιρεία συμφωνούν με την ε, δήλωση προέλευσης, τότε αυτό που κάνουμε είναι να διεξάγουμε ελέγχους στο εργοστάσιο και ε, να εξετάσουμε το κάθε εξάρτημα για να διαπιστώσουμε την προέλευσή του. Και γι' αυτό διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Όταν ξεκινάς δηλαδή από μια χώρα και καταλήγεις μέσα από πολύ μεγάλες δρομές σε μια άλλη, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και τι σημαίνει αυτό, λέει ο Πρόεδρος, για το μέλλον. θα υπάρξει μια εναλλακτική, θα υπάρξει μια λύση ή θα μείνει τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως είπα στην ε, παρουσίαση, για παράδειγμα, κανόνες πολύ πιο ευέλικτοι σε σχέση με το 2011, που χρησιμοποιούνται ήδη και οι εξαγωγείς από τις τρίτε χώρες του χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο από τους δικούς μας φορείς. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές από την Κορέα. Δεν έχω τα ακριβή ποσοστά, αλλά το 90% των εξαγωγών από την Κορέα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποφελούνται από, αυτές τις, ε, από αυτούς τους προτιμησιακούς ε, δασμούς. Αντίστοιχα, το 75% των δικών μας εξαγωγών προς την Κορέα υποφελείται από τις ίδιες ε, προτιμήσεις. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, ε, έγινε και αυτή η έρευνα από εμάς πέρυσι, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις ανάγκες και να προσαρμοστούμε βελτιώνοντας το πλαίσιο. Επίσης, όταν βλέπουμε τους ε, εταίρους μας από τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν τους δικούς μας κανόνες κατά 90% ή και περισσότερο 100%, τότε νομίζω πως μάλλον κάτι έχουμε κάνει σωστά. Μαζί με την Ορβηγία και τον Καναδά, οι δικοί μας κανόνες ε, θεωρούνται από τους καλύτερους, διότι βοηθούν τους δικούς μας φορείς να τους ε, χρησιμοποιήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο όφελος αλλά και μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Ωραία λοιπόν, θα σας εξετάσω συνάδελφοι να το γνωρίζετε. Ευχαριστούμε. Σημείο 16. Έκθεση για την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε συζητήσει επί μακρόν την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες, στην ε, Ιορδανία, στη Μολδαβία και σε άλλες, ιδιαίτερα στην Ουκρανία. το 2018 εγκρίθηκε το τέταρτο μέσο χρηματοδότησης και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης συζήτησης ήταν η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για, το δεύτερο κομμάτι χρηματοδότησης προς την Ουκρανία. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να συζητήσουμε για την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ουκρανίας. Μαζί μου είναι ένας εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ, ο Σαντιάγο Λοράντζα Γκαρσία, ο οποίος θα μας ενημερώσει για περίπου 5-7 λεπτά για την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Λάγκη, και καλησπέρα σε όλους σας. Είναι χαρά για μας να σας βλέπω σε αυτή τη νέα θητεία, στη νέα νομοθετική περίοδο και χαίρομαι που σας βλέπω όλους ως μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παρουσιάσουμε σήμερα την έκθεση για τη μακροοικονομική συνδρομή. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό πέρσι και χαίρομαι που μας δίνετε αυτή ε, την ευκαιρία. Ε, δεν ξέρω αν ξέρουν όλα τα μέλη τι είναι η μακροοικονομική βοήθεια. Και επίσης ε, θα σας, κάνω και ένα, θα σας δώσω ένα στιγμιότυπο των ε, Δύο λόγια για το ε, μακροοικονομικό μέσο. Δεν είναι ένα τυχαίο εργαλείο, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να δώσει βοήθεια μόνο σε χώρες εταίρους ε, και θέλουν να καλύψουν χρηματοοικονομικά κενά ως τμήμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί μόνο αναπερίπτωση όταν υπάρχει περίπτωση κρίσης. και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα συνήθη προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ε, ιδέα είναι να δούμε την μακροοικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε οικονομικές προσαρμογές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βάλουν τα κράτη σε μία βιώσιμη οδό. Και επίσης ε, πρέπει να είναι ε, και κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει χώρες οι οποίες είναι υπερχρεωμένες. Και φυσικά είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνεται υπό όρους. Υπάρχουν όροι με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν χώρες δικαιούχοι που πρέπει να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς και ε, δίνεται σε δόσεις. Οι δόσεις εξαρτώνται ε, από μια σειρά από διαρθρωτικά ε, μέτρα μεταρρυθμίσεων, συμφωνούνται με τη χώρα και έχουν τη μορφή μνημονίου συνεννόησης. Και υπάρχει και ένας τρίτος τύπος ε, αιρεσιμότητας, συνδέεται και με ένα πρόγραμμα προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Uh, uh, e- Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση από τη συνήθεια ευρωπαϊκή ε, συνδρομή συνεργασίας που είναι ε, αυτό το οποίο δίνεται συνήθως. Ε, τώρα, τι καταφέραμε το 2018 και την αρχή του 2019. Καταρχάς, ε, το 2019 18 συγγνώμη, εγκρίθηκαν δύο αποφάσεις, ε, το μακροοικονομικό μέσο για τη Γεωργία και 2 ε, δις ευρώ και την, στη Γεωργία 1,4 δις ευρώ αντιστοίχως. Και για τις δύο χώρες αυτές έχει ήδη εκταμιευθεί η πρώτη δόση. Για την Ουκρανία, η Ουκρανία κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις για την πρώτη δόση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να εκταμιεύσει τον Δεκέμβριο του 2018 τη δόση αυτή. Ε, δόθηκε και ένα ενημερωτικό σημείωμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας όλες τις λεπτομέρειες ε, για την αιτιολόγηση, για το ε, πώς θεωρούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τώρα, μετά... Ε, είχαμε και προεδρικές εκλογές ε, και αυτό σημαίνει ότι καθυστέρησε λίγο η τήρηση κάποιων προϋποθέσεων. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση τώρα στην Ουκρανία και θεωρούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις προϋποθέσεις. Ε, τώρα για τη Γεωργία. Η πρώτη δόση εκταμιεύτηκε, ε, ήταν 30 εκατομμύρια και υπάρχουν ακόμα 25 διαθέσιμα. Αυτό δεν συνδέεται. Η πρώτη δόση δεν συνδεόταν με προϋποθέσεις και οι γεωργιανές αρχές κατά την άποψή μας έχουν προχωρήσει ε, ε, στις εφαρμογές αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ίσως πριν το τέλος του έτους ε, να ε, έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Σε θέματα ανατολική γειτονία υπάρχει και ένα τρίτο πρόγραμμα για τη δημοκρατία της ε, Μολδαβίας. Είναι ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια μεικτή επιχείρηση που περιλαμβάνει επιδοτήσεις και δάνεια και τα κονδύλια είναι διαθέσιμα μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Η πρώτη δόση, τα 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι σε αναμονή γιατί οι πολιτικές προϋποθέσεις δεν θεωρείται ότι έχουν καλυφθεί ακόμα. Αυτό οφείλεται σε διάφορες ε, ανησυχητικές τάσεις που περιελάμβανε και την ακύρωση των ε, δημαρχικών εκλογών ε, στο Τσιθινάου το 2018 και ε, υπάρχουν διάφορες σοβαρές δημοκρατικές οπισθοχωρήσεις στη Μολδαβία αυτή τη στιγμή. Μετά, τον Ιούνιο του 2019 ανέλαβε νέα κυβέρνηση και εδώ δόθηκε μια νέα δυναμική και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει πρόγραμμα και, ε, και αυτό έχει αναστείλει την εφαρμογή του ε, εν αναμονή των εξελίσεων. Ε, τελικά είχαμε μία συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού που είναι το πρώτο επιτυχές στάδιο και μετά από όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις αναμένουμε να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε τελικά την πρώτη και ίσως και τη δεύτερη δόση εντός του 2019. Ε, ήρθαμε αμέσως σε επαφή με τις αρχές της Μολδαβίας και τη νέα κυβέρνηση και ε, βλέπουμε πού ακριβώς βρίσκονται για να δούμε πού μπορούν να, να υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ε, στην ε, τήρηση των υποχρεώσεων, ώστε να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε με ασφάλεια. Τέλος, υπάρχουν και δύο ακόμα ε, ενεξελίξει διαδικασίες στη νότια γειτονία. Η μία είναι η Ορδανία, η οποία ολοκληρώθηκε. Είχαμε μία πλήρη επιχείρηση 200 εκατομμυρίων ευρώ και η δεύτερη και τελευταία δόση έγινε εντό του 2019. Και επίσης έχουμε μία ε, επιχείρηση σε εξέλιξη ακόμα στην Τινησία. Το συνολικό ποσό είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και εκρεμεί ακόμα η τελευταία τρίτη δόση 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, και πάλι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις αρχές ε, ώστε να ε, βεβαιωθούμε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Να πω δύο λόγια τώρα για τις μελλοντικέ επιχειρήσεις και τις προπτικές του ταμείου αυτού, του μέσου αυτού. Αυτή τη στιγμή στα Σκαριά υπάρχει μόνο μία επιχείρηση για την Ιορδανία. Η Ιορδανία έστειλε επιστολή ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράταση του μακροοικονομικού μέσου για 500 εκατομμύρια ευρώ ε, και αυτό είναι τμήμα μιας ε, ε, γενικότερης παγκόσμιας επιχείρησης διεθνούς στήριξης η οποία είχε ξεκινήσει με μια διάσκεψη στο Λονδίνο στις αρχές του έτου και έχετε και σε συνέχεια μια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εάν ε, είχε πλήρη επιτυχία το προηγούμενο μακροοικονομικό μέσο να ε, εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να υποβάλει πρόταση τις επόμενες εβδομάδες και φυσικά προσβλέπουμε να τα συζητήσουμε μαζί σας και φυσικά να τα παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει με τη μακροοικονομική συνδρομή στα πλαίσια του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Μάιο πέρσι μια πρόταση για τον επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και μεταξύ των προτάσεων ήταν και η δημιουργία ενός νέου μέσου, το λεγόμενο NDG, ε, μέσω ε, ανάπτυξης γειτονίας και διεθνούς συνεργασίας. Αυτό θα συνενώσει διάφορα προγράμματα και μέσα για να μπορέσουν ε, να ε, συντονιστούν. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το μακροοικονομικό μέσο έχει διακριτά χαρακτηριστικά που σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει ως ξεχωριστό μέσο στο μέλλον. Ε, βεβαίως ε, απαιτείται πολύ στενός ε, στεντονισμός με το νέο μέσο το NDG, αλλά οι επιχειρήσεις ε, για το μακροοικονομικό μέσο θα ενεργοποιούνται ad hoc με βάση αποφάσεις οι οποίες θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διαδικασία της συναπόφασης. Με αυτό ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το στιγμιότυπο. Όπως σας είπα, το μακροοικονομικό μέσο είναι μέσο επίγουσας ανάγκης και η αποτελεσματικότητα της απόφασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ε, από τη στενή συνεργασία μεταξύ των συνομοθετών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα την Επιτροπή τη δική σας. Ε, όπως σας είπα λοιπόν, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και στις ε, συζητήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως ώστε να εγκρίνονται σύντομα οι προτάσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ε, Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και ιδιαίτερα για το πρώτο τμήμα που μας εξηγήσατε τη μακροοικονομική βοήθεια. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Η κυρία Ροντρίγκε Πινέιρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Εγώ την περασμένη θητεία μου είναι συγγήτρια των σοσιαλιστών για τη μακροοικονομική βοήθεια στις γειτονικέ χώρες. Μεταξύ αυτών ήταν και η Γεωργία. Και προφανώς είμαι μεγάλη υπέρμαχος αυτού του μέσου, γιατί είναι πολύτιμο για να βοηθήσει αυτές τις χώρες να προχωρήσουν προς τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στηριχθούν. Είναι γεγονός ότι στη Γεωργία είδαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές ε, και στα θέματα του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Αλλά φυσικά απομένει ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσει στους στόχους της υγειοργίας, στους στόχους που θέσαμε από κοινού. Θα ήθελα όμως ιδιαίτερα να σας ρωτήσω τα εξή τρία συγκεκριμένα. Είπατε πρώτα απ' όλα ότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτεμευτεί και η τελευταία δόση των 30 εκατομμυρίων. Τι εκκρεμεί ακόμα, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Γεωργία για να ε, πληρωθούν τα κριτήρια του μνημονίου. Ε, δεύτερον, έχω την αίσθηση ότι για να αναπτυχθεί βιώσιμα η Γεωργία πρέπει να αληθεί το θέμα ε, της έλλειψης κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού. Αυτό πώς προχωράει. Και το θέμα της πρόσβασης στη γη. Και αυτό είναι από τα βασικά θέματα που φάνηκαν από τα σημαντικότερα ε, όταν χρειάστηκε βοήθεια για να παραμείνει εκεί ο πληθυσμός και να μειωθούν οι ανισορροπίες οι εδαφικές που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Και δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το θέμα σήμερα. Και τέλος, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που προβλέπονται για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορούν να επωφεληθούν από τη συμφωνία. Πώς έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ ο Χέλμοντ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Γιατί η έκθεση ήταν αρκετά συγκεκριμένη και ακριβής. Ωστόσο, μιλώντας για την Ουκρανία, είπατε ότι ε, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα κριτήρια για τη μακροοικονομική βοήθεια για να εκταμιευθούν τα χρήματα. Ερώτηση λοιπόν και κοιτάω και τα στοιχεία. Το 2019 με τη νέα κυβέρνηση καταβλήθη πραγματικά μια προσπάθεια κατάδειξης ε, της πολιτικής βούλησης για να γίνουν επιπλέον μεταρρυθμίσεις με τρόπο ώστε να θεωρηθεί αυτό ικανοποιητικό. Δόθηκαν όμως τα χρήματα πριν αυτή την τελική φάση με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, για τη διαφάνεια κτλ. Έχουν αρχίσει όλα αυτά, αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς είμαστε τόσο σίγουροι ότι τα χρήματα που δίνουμε στην Ουκρανία έπιασαν τόπο και βοήθησαν για να βελτιωθεί η πολιτική, νομική, οικονομική κατάσταση στη χώρα. Γιατί παραμένει η ψαλίδα ανοιχτή στη χώρα και στις κοινωνικές προδιαγραφές και μάλιστα ανοίγει ακόμα περισσότερο. Πώς βεβαιωνόμαστε λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά που εκταμιεύουμε και συνδέονται με προϋποθέσεις πιάνουν τόπο και φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους και εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Άλλη ερώτηση για τη Μολδαβία τώρα. Γνωρίζουμε ότι με τη νέα κυβέρνηση έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ήρθε και ο Πρωθυπουργό ή Πρωθυπουργό μάλλον ε, τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο και ζήτησε την υποστήριξή μα. για να επιστρέψουν κάποια χρήματα που είχαν φύγει με ένα τραπεζικό σκάνδαλο. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια νομίζω. χάθηκαν τα χρήματα, τα σταμάτησα τα, ε, και εμείς δεν, δεν τα δικά μας. Ε, θα βοηθήσουμε να ορθοποδήσει η χώρα με τη νέα κυβέρνηση. για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από τα προαπαιτούμενα και τους όρους που βάζει η χρηματοοικονομική ε, βοήθεια αυτή, η μακροοικονομική καλύτερα. Είναι λίγο φαύλος κύκλος. Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Όχι μόνο εμείς στη δική μας Επιτροπή, αλλά γενικότερα το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω για την, την Ισία. Έχετε κανένα νέο από εκείνο το μέτωπο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχω και αναπληρωτή, τον Τζον Γκρίς, ο οποίος θα σας μιλήσει γιατί ειδικεύεται ιδιαίτερα σε θέματα Ουκρανίας και Γεωργίας. Να απαντήσω για τα δύο τελευταία, για τη Μολδαβία και την Τινησία. Φυσικά η Μολδαβία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτό ήταν και αντικείμενο για μεγάλη ανησυχία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί, ε, ως θεσμικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε υποστηρίξει πάρα πολύ τη νέα κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί και προσπαθούμε και εμεί να τους βοηθήσουμε. Έχουν ενστενιστεί πλήρω τι μεταρρυθμίσει. είναι κτήμα πια ε, ε αυτές που αναφέρονται στο μνημόνιο της μακροοικονομικής βοήθειας ε, θέλουν να τις υποστηρίξουν θέλουμε και εμείς να τις υποστηρίξουμε για να τις εφαρμόσουν ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά η ίδια η κυβέρνηση πραγματικά ε, τις θεωρεί κτήμα της. Έχει την ιδιοκτησία όπως λέμε. Και από αυτές θα εξαρτηθεί και η επιτυχία της στρατηγικής για την ανάκτηση ε, των χαμένων των χρημάτων που χάθηκαν από το σκάνδαλο το τραπεζικό. Και έχει αναλάβει γρήγορη δράση εδώ η κυβέρνηση της Μολδαβίας. Χρειάζονται υποστήριξη. Ζήτησαν υποστήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι θα υποστηριχθούν και από τους δύο. Έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για να εκταμιευθούν οι πρώτες ε, δόσεις. Υπάρχουν για τη δεύτερη και την τρίτη δόση κάποιες άλλες προϋποθέσεις που είναι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα. Τις συζητούν τώρα και τις προωθούν. Πάντως γενικά, παρόλο που είναι πολύ φιλόδοξες οι μεταρρυθμίσεις, είμαστε σε καλό δρόμο και ευτυχώς και πάλι θα είμαστε σε θέση πριν τα τέλη του έτους να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της δεύτερης δόσης. Την Ισία. Δεν είναι εύκολη χώρα η Τινησία. Υπό ποια έννοια. Δεν ήταν καθόλου εύκολος ο δρόμος για τους ίδιους να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Είναι και η πολιτική κατάσταση και η δυσκερής για να πάρει κανείς δύσκολα μέτρα. Και στα οικονομικά, ορισμένα από τα μέτρα, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με το δούνο του, δεν ήταν καθόλου εύκολα στη λήψη τους. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν βελτιώνεται ουσιαστικά η κατάσταση. Και η έλλειψη αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ένας από τους λόγους που δεν προχωρούν. Έχει συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό, κάνουν πρόοδο η Τινησή, αλλά και πάλι πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ κοντά στην εκταμίευση. Το επόμενο δίμηνο ε, μπορούμε φαντάζομαι να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της τρίτης και τελευταίας δόσης. Για το μέλλον η Τινησία ίσως να είναι μία από τις χώρες που θα μας τυπήσει την πόρτα για να ζητήσει και νέα βοήθεια σε περίπτωση που ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρούσα. Είναι μεγάλες οι οικονομικές ανάγκες και χρειάζεται η χώρα και θα χρειαστεί τη διεθνή υποστήριξη ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις εξελίξεις και τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. Λοιπόν, για τη γεωργία καταρχάς. Όντως συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές της χώρας έτσι ώστε να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις Φυσικά αυτό γίνεται σταδιακά, υπάρχει ανάληψη ευθυνών. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ε, προϋποθέσεις οι οποίες ε, ακόμα παραμένουν ανοιχτές, όπως για παράδειγμα η ασφάλιση ευθύνης τρίτου μέρους. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων, των οχημάτων. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτό το τομέα μια κάποια εναρμόνιση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και ένα προαπαιτούμενο για την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση της αγοράς στη Γεωργία. Βέβαια αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και δεν είναι κάτι εύκολο να κάνει άλλωστε η κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εκκρεμότητα επίσης. Η κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ένα, νομο, ένα σχέδιο νόμου για την εταιρική νομοθεσία όπου θα ρυθμίζονται οι μορφές των εταιριών, θα υπάρχει κάποια προσέγγιση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο να μπορούν να συγκριθούν με ε, τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Στη Γεωργία δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια προς το παρόν σε ό,τι αφορά τη μορφή των εταιριών. Επίσης, το νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον των ε, φορέων της ε, χώρας και υπάρχει κάποια βούληση για πρόοδο. Μέσα στο μήνα θα έχουμε νεότερα. Για ορισμένες από τις άλλες προϋποθέσεις, ε, για παράδειγμα τη στρατηγική για την αγορά εργασίας, να σας πω ότι έχει γίνει μια διαβούλευση, έχει περάσει αρκετός καιρός και είναι καλό αυτό, διότι πάντα είναι σημαντικό να ακούμε και τη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Μετά, αν κατάλαβα καλά, κάνατε μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με την εκπαίδευση και την ε, μεταρρύθμιση στην, στην Ήπεθρο. Υπάρχει σχετική νομοθεσία. Πρόσφατα ψηφίστηκε ε, νόμος για την εκπαίδευση και κατάρτιση, ο οποίος αποτελεί πλαίσιο για τον ε, τομέα αυτόν και επίσης δίνει τη δυνατότητα σε διάφορες ενισχυμένες μορφές συνεργασίας και σε μακροοικονομική συνδρομή. Μετά, το θέμα της ε, αγοράς γης. Υπήρξε ένα θέμα ακτιματογράφησης. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τις αρχές ε, για να απλουστευτεί η διαδικασία καταγραφής και ακτιματογράφησης. Υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια 300.000 περίπου που πρόκειται να ακτιματογραφηθούν. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει αυτό το ορόσημο η Γεωργία και οι αρχές της χώρας τώρα προσπαθούν, όπως σας είπα, να απλουστεύσουν τη διαδικασία εκτιματογράφησης και σε δεύτερο στάδιο θα γίνει και μηχανογράφηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κίνητρα για να γίνει εθελοντικά αυτή η διαδικασία από τους ε, κατοχούς γης. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο συστηματικής ε, καταγραφής και στο τέλος θα, έχει, θα έχουν καταφέρει να εναρμονιστούν πλήρως. Τώρα, για την πρώτη δόση. Ε, το Νοέμβριο του 2018 η κυβέρνηση κατάφερε να πιάσει τους στόχους η κυβέρνηση της Ουκρανίας, για την Ουκρανία μιλάμε και έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις από τις αρχές, ε, έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα Ο κοινωνικός ε, τομέας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, διότι σε μία περίοδο οικονομικής χρήσης, όταν μια χώρα δεν λαμβάνει εξωτερική βοήθεια, η προσαρμογή πρέπει να γίνει με πιο απότομο τρόπο. Ένα ε, τρόπο ο οποίος θα είναι πιο επώδυνος για τους πολίτες. Έπειτα. Υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την μακροοικονομική συνδρομή, για παράδειγμα ένα σχέδιο βοήθεια στα νοικοκυριά, το οποίο είχε ως στόχο να καλύψει την αύξηση στην τιμή του αερίου. Αυτή ήταν και μία προϋπόθεση για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, ε, η οποία πλέον έχει πραγματοποιηθεί. Και να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Σαντιάκο, το μακροοικονομικό μέσο δεν προορίζεται για εκείνους τους μεμονωμένους πολίτες που έχουν ανάγκη τα χρήματα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο θα ε, χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση της Ουκρανίας έτσι ώστε να στρώσει το έδαφος ε, για βελτιώσεις, για μεταρρυθμίσεις, για περισσότερες κοινωνικές ε, δαπάνες. Χρηματοδοτούμε δηλαδή την κυβέρνηση Ουκρανίας για να πραγματοποιήσει αυτές τις αλλαγές. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κάνιας έχει μία ακόμα ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσφάτως ο νυν υπουργό Εξωτερικών και μέλλον υπάτος εκπρόσωπος, ο κύριος Μπορέλ, είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ενίσχυση προς, την, προς το Μαρόκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τη διακίνηση ανθρώπων και τη ε, διακίνηση ναρκωτικών παράνομων ουσιών ε, στα ε, σύνορά μας με τη Βόρεια Αφρική επειδή χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός μακροοικονομικής βοήθειας ad hoc με κάποιες χώρες, θα μπορούσε ίσως να είναι και ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, κατόπιν αιτήματο του Βασιλείου του Μαρόκου, για παράδειγμα, για να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στα βόρεια της χώρα ώστε να έχουμε καλύτερη ε, έλεγχο των ε, ροών παράνομων μεταναστών και παράνομων ουσιών. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι. Για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι ευτυχώ για το Μαρόκο έχουν ε, σχετικά καλή οικονομική κατάσταση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες και τις παραμέτρους, ιδίω ε, ε, ο εξωτερικός κλάδος ε, είναι σε καλή κατάσταση, επομένως δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία χωρών που έχουν αδυναμίες στον εξωτερικό τομέα και ιδιαίτερε χρηματοοικονομικές ανάγκες και να χρειάζονται χρηματοοικονομική προσαρμογή. Και επειδή ακριβώς ε, έχει έτσι κατάσταση, το Μαρόκο δεν έχει πρόγραμμα ε, προσαρμογής ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι προϋπόθεση. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά για να βρίσκονται με τη σωστή πλευρά των οικονομικών πολιτικών, να έχουν εύρωστες οικονομικές πολιτικές, αλλά δεν είναι πρόγραμμα χρηματοδότησης, επομένως δεν είναι επιλέξιμο αυτή τη στιγμή για μακροοικονομική συνδρομή. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 17 είναι τα διάφορα, το είναι το αγαπημένο μου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Το 18 είναι η επόμενη συνεδρίασή μας, 23 και 24 ε, Σεπτεμβρίου. Σύντομα λοιπόν. Και με αυτό ολοκληρώνεται η συνήθη συνεδρίαση, η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας για σήμερα και θα ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά με τη συνεδρίαση των συντονιστών της ε, Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Ένα διάλειμμα λοιπόν 5 λεπτών.